Δεν αναφέρεται πια ε, τοποθέτηση σε ό,τι αφορά της έρευνα ε, της Όλαφ βάση τη 173 του 99 και του κανονισμού γρατόμ ε, του 1999. Την τοποθέτηση αυτή λοιπόν την έλαβα και Ο τίτλος ε, αναφέρεται και στα πρακτικά της συνεδρίασης. Ε, διατίθεται ε, από αύριο για τρεις μήνες μέχρι από 15 Μαρτίου δηλαδή 2013 και περνάμε σε συζήτηση για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία ώρα διαρκούν τα, οι συζητήσεις αυτές. Πρώτο θέμα η συζήτηση για το, την κατάσταση των Μπαγκλαντές. Το λόγο έχει καταρχάς ο συνάδελφος Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ήμουν στην Τάκα, πριν από πέντε χρόνια επισκέφθηκα το Εθνικό Μουσείο Απελευθέρωσης και διαπίστωσα τις φρικαλαιότητες που διαπράχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1971 για την ανεξαρτησία. Πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο και τέσσερις δεκαετίες έχουν περάσει, αλλά υπάρχει ατιμορρησία για τους εγκληματίες πολέμου. Είναι αδικαιολόγητο το να μην επιτρέπεται να δικαστούν μέσα σε ένα πλαίσιο κατάλληλης διαδικασίας για τέτοιου είδου εγκλήματα κανένα καθεστώ περιορισμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται. Και επίση δεν είναι λογικό να ζητήσουμε από του Μπαγκλαντεσιανού να του δικάσουν ε, ε, στο εξωτερικό εκτό τη δικαιοδοσία του. Γι' αυτό θα πρέπει να καταδικάσουμε την πρόσφατη βία που εμπνέεται από τον Τζαμάλ Ισλάμι και πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση ώστε να επικρατήσει τάξη και οι ετοιμιγορίες αυτών των δικών να φέρουν τέλος σε αυτή την τρομερή περίοδο της ιστορίας της χώρας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Τάνο και τώρα για δύο λεπτά στον Αλφός Μπρέντα. Ευχαριστώ. Μια και εγώ ανέλαβα την πρωτοβουλία και ζήτησα να συμπεριληφθεί στα κατεπήγοντα σήμερα τον Μπαγκλαντές, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να αντιδράσουμε άμεσα σχολιάζοντας ε, την ε, θανατική καταδίκη του Αντιπροέδρου του κόμματος ΑΜΠΑΚ. Δεν μπορούμε να, να αγνοούμε τόσο σημαντικά πολιτικά γεγονότα στο Μπαγκλαντές. Και είναι ε, παράδοξο το θέμα ότι ε, το Δικαστήριο ε, Εγκλημάτων Διεθνούς Δικαίου θα πρέπει να βοηθήσει τον Μπαγκλαντές να γυρίσει σελίδα στην ιστορία του μετά τον πόλεμο του 1971. Φυσικά θα πρέπει να καταδικάσουμε τη θανατική ποινή και να ζητήσουμε τη μετατροπή των θανατικών καταδικών και την θέσπιση μορατόριου για τις θανατικές ποινές. Επίσης θα πρέπει να τηρηθούν ε, τα εχέγγυα της δίκης δίκης. Ε, είναι απαραίτητο κάτι ιδιαίτερα για ένα δικαστήριο που θα πρέπει να προωθήσει την εθνική συμφιλίωση. Μάλιστα, οι βιοπραγίες που ακολούθησαν την ε, έκδοση των αποφάσεων είναι απαράδεκτες. Ε, διαπράχθηκαν και από, τους, από τα μέλη της Τζαμάτ, αλλά και από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ε, η ειρηνική διαδήλωση είναι θεμελιώδης ε, δικαίωμα και η βία σε καμία περίπτωση δεν είναι μια λογική απάντηση σε τέτοια φιλοειρηνική διαδήλωση. Είναι ανησυχητικό το στοιχείο και η πληροφορία της Human Rights Watch ότι τα περισσότερα θύματα είναι θύματα των δυνάμεων ασφαλείας ε, της αστυνομίας του Μπαγκλαντές. Άλλωστε, τα πρόσφατα επεισόδια βίας δείχνουν την πόλωση της κοινωνίας των Μπαγκλαντές και την αντιπαράθεση του κοσμικού στοιχείου με το θρησκευτικό που εκπροσωπεί το Εθνικό Κόμμα του Μπαγκλαντές. Με το ψήφισμά μας απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα κόμματα για να υπερβούν τις διαφορές τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Πρέντα. Και τώρα Ευχαριστώ. Μετά την ε, έκδοση της 5 Φεβρουαρίου της ε, ε, καταδίκη σε θανατική ποινή του κυρίου Σαΐντι δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα και διαταραχές στον Μπαγκλα... Βέβαια ο, ο κατα... κατηγορείται για σημαντικά εγκλήματα πολέμου, βιασμούς, δολοφονίες μην ξεχνάμε ότι 300.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και είχαμε και πολλούς ε, ε, θανάτους. Και είχαμε και, σε επεισόδια αυτά όμως ε, μετά τις διαδηλώσεις είχαμε τραυματισμούς πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε αυτή την έκδοση θανατικών καταδικών. Είναι από τις λίγες χώρες που έχουν, εφαρμόζουν τέτοιες θανατικές ποινές. Θα πρέπει να ξυλιτεύσουμε αυτή την έκδοση θανατικής καταδίκης που δεν δικαιολογείται από τα διαπραχθέντα εγκλήματα. Γι' αυτό ζητούμε πάγωμα της θανατικής ποινής και ζητούμε από το Μπαγκλαντές να επανέλθει στο σεβασμό των διεθνών προδιαγραφών σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. 1,5 λεπτός η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ πρόεδρε και μιλώ και ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας για την Νότια Ασία και ως, μέτρος, ως μέλος του Κούβια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σε ό,τι αφορά τα θέματα των ε, ε, βιοπραγιών που έχουν λάβει χώρα ε, τα τελευταία 40 χρόνια την δράση του δικαστηρίου η δέσμευση για τις δίκες αυτές ήταν μέρος του μανιφέστο στις τελευταίες γελικές εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων έγινε ευρέως αποδεκτό και πλέον το κόμμα αυτό είναι στην κυβέρνηση. Νομίζω όμως ότι πολλοί έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα σε ό,τι αφορά στο θέμα αυτό αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν αυτέ οι δίκε, αλλά αποδοκιμάζουμε το γεγονό ότι συμπεριλαμβάνονται ακόμα οι θανατικέ καταδίκες. Κατανοούμε την πολιτική διάσταση ε, τη δίκη αυτή, αλλά θεωρούμε ότι τα δικαστηρία θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητα και ότι η πολιτική ανάμειξη από οποιοδήποτε ε, μέτωπο θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα αναφέρεται απαράδεκτο. Καταλαούμε την επιθυμία των παγκλαντές να ε, επεξεργαστεί το παρελθόν του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μην τηρούνται τα διεθνή πρότυπα. Και πλέον υπάρχουν ανησυχίε σε ό,τι αφορά την, ε, το δικαίωμα ανταγωγή κτλ. Και καταλαβαίνουμε φυσικά ότι προκαλούνται έντονα συναισθήματα, αλλά όπως έχουμε πλέον πολλοί μαρτύρες να μας ε, μαρτυρήσουν, ότι, υπάρχει, ότι είναι αρκετά τόσο ο θάνατος και βιοπραγίες και στο στόχαστρο είναι συχνά οι μειονότητες ε, με την ε, χρήση πυρομαχικών κατά των ε, πολιτών. Καλούμε λοιπόν προς όλες, από όλες τις, όλες τις πλευρές να σταματήσουν τη βία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λάμπερτ. Ένα λεπτό, η κυρία Βίξτρομ. Det är av utomordentlig vikt att alla de människor som σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τα όσα συνέβησαν από το 1978 και είναι απόλυτα λογικό ένας υπεύθυνο για γενοκτονία να πρέπει να λογοδοτήσει. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ποινές που επιβάλλονται να είναι ισότιμες και να δισεύονται οι δικαστικές διαδικασίες στο δικαίωμα στην ε, υπεράσπιση. Αυτή τη στιγμή όμως, μέχρι μάλλον σήμερα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο κατάλογος των παραβάσεων του δικαίου του και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ μακρύς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απαχθεί πριν από την δίκη, άνθρωποι οι οποίοι περάσαν ακροματική διαδικασία χωρίς ε, βοήθεια δικαστική και ακόμα κι αν Θεωρούμε ότι είναι ένοχοι. Οι δίκες θα πρέπει να είναι δίκαιες και γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει και να ζητήσει από τον Παγκλαντές να θέσει τέλος σε αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Κυρία Βεριζιά τώρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 1971 ο πόλεμος της ανεξαρτησίας ε, μεταξύ του Ανατολικού και του τότε Δυτικού Πακιστάν οδήγησε σε χιλιάδες για να μην πούμε εκατομμύρια θύματα. Φυσικά ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θύματα και να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Το 2010 συστήθηκε ένα δικαστήριο για να ε, εκδικάσει τέτοιου είδους εγκλήματα διεθνούς δικαίου. Βέβαια, η αποφάση αυτού του δικαστηρίου ε, δημιούργησε μια έξαρση της βίας. Δεν μπορεί ε, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να παραβιάζει τους διεθνούς ε, κανόνες και περιοδιαγραφές και ιδιαίτερα το δικαίωμα για μια δίκη. δίκη. Δεν μπορεί να τροποποιεί την νομοθεσία για το δικαστήριο αυτό μετά τις πιέσεις του κόσμου, ούτε να, να ενδίδει σε τέτοιες πιέσεις. Αυτό δυστυχώ συνέβη. Είχαμε καταπιέσει καταστολή και η κυβέρνηση μαζί με τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να επαναφέρουν την τάξη, για να αποφύγουμε επανάληψη των αποτροπιαστικών και αποτρόπαιων ενεργειών. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Τώρα ξεκινούμε με τον κύριο Κατσμάρεκ από τι πολιτικέ ομάδε Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. κυρίε και κύριοι. Ε, σίγουρα είναι δικαιολογημένη και εύλογη η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνη. Ε, πολλό δε μάλλον ε, όπω στον Παγκλαντές ε, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τη διάπραξη των εγκλημάτων, αλλά δεν θα πρέπει στο όνομα της δικαιοσύνη να οδηγούμαστε σε νέε παραβιάσει του δικαίου και σε βιοπραγίες. Τέτοιου είδου φαινόμενα θα πρέπει να τα, να τα αποφύγουμε. Η επανένωση και η συμφιλίωση αλλά και η απονομή τη δικαιοσύνη θα είναι ευκολότερες αν ε, δεν εφαρμοστούν οι θανατικές ποινές. Δικαίως ε, ε, απαιτούμε στο ψήφισμα να γίνουν πιο ήπιες οι ποινές, να καταργηθεί η θανατική ποινή και να εφαρμοστεί στο μεταξύ ένα μορατόριο. Θα πρέπει επίση να τηρηθούν οι αρχέ τη ανεξιθρησκεία, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην γίνει προσφυγή στη χρήση βία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε τώρα ένα λεπτό η κυρία Κρέτου. Σας ευχαριστώ. Εδώ και πολύ καιρό ανησυχούμε από τις, ε, τη διαθρησκευτική βία στον Μπαγκλαντές. Κατανοούμε την ανάγκη ε, για δικαιοσύνη, αλλά ε, όπως είπε και το Ευρωκοινοβούλιο επαναλημμένως, η θανατική ποινή δεν μπορεί να είναι δίκαιη. το, η τιμωρία ενός εγκλήματος μέσω ενός άλλου εγκλήματος δεν μπορεί παρά να επιτείνει τις εντάσεις στη χώρα. Ζητάμε από τις αρχές να παγώσει την θανατική ποινή των υπευθύνων για τις ε, αποτρόπες πράξεις του 78. Ε, Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφευθούν ευθύ η βία όπως στις τελευταίες εβδομάδες η βία ποτέ δεν είναι η λύση η κυβέρνηση πρέπει να επιμείνει και να ε, επικρατήσει ένα κλίμα ειρηνευτικό Ευχαριστώ σας ευχαριστώ και τώρα ένα λεπτό ο συνάδελφος Μπενιόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ακούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τόσο στο Κοινοβούλιο έχουμε καλές σχέσεις με το Παγκλαντές και με τη διασπορά του Παγκλαντές και με... συνεργαζόμαστε και με τις σχετικές υπηρεσίες και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε και δικαίωμα και καθήκον να μιλήσουμε η χειρά για αυτά που μαρτυρούμε, την πρόσφατη βία την οποία την προκάλεσε η έλλειψη εμπιστοσύνης γιατί οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου και οι αναφορές ε, για πολιτική ανάμειξη στο Διεθνές Δικαστήριο έχουν γίνει τόσο πασίφανείς που πρέπει να παρέμβουμε. Καλό και εγώ για μορατόριο μου στην θανατική καταδίκη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να ζητήσει διεθνή αρρωγή σε ό,τι αφορά και το πεδίο εφαρμογής από πλευράς του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός ειδικού διεθνούς δικαστηρίου για να υπάρχει εμπιστοσύνη σε δίκαιες δίκες να είναι βέβαιη όλη η κοινωνία για τα αποτελέσματα και το, τις δικαστικές αποφάσεις προκειμένου να είναι βέβαιοι όλοι ότι θα τιμωρηθούν οι υπέτοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο συνάδελφο Μπιέλαν, ένα λεπτό. Η κατάσταση των Μπαγκλατές ήταν ήδη περίπλοκη και τις τελευταίες εβδομάδες έχει επιδεινωθεί. Ήταν δίκαιη και εύλογη η ανάγκη απόδοσης της δικαιοσύνης, αλλά η οι διαδηλώσει δείχνουν ε, την πόλωση της ε, Μπαγκλαντισιανής κοινωνία μετά από τέσσερι δεκαετίες ε, από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Δυστυχώς η Ινδουιστική μειονότητα υπόκειται σε διώξεις, 40 ιερά έχουν καταστραφεί, γίνονται ληστείες ή εμπρισμοί σε καταστήματα Ινδουιστών φαίνεται ότι η πόλωση οφείλεται σε θρησκευτικού λόγου. Η ανάγκη επαναφορά τη ε, δικαιοσύνη και τη επανασυμφιλίωση θα πρέπει να συνοδευτεί με έκκληση προ τι παγκλατισενές αρχέ να επανέλθουν στο δρόμο του δικαίου και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς προδιαγραφές. Μόνο τότε το Δικαστήριο Εγκλημάτων Διεθνούς Δικαίου θα ε, διαδραματίσει το ρόλο του. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η διαφάνειά του και να αποκατασταθεί η τάξη σε μια κοινωνία που απειλείται από τα ταραχές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαστάλκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το προτινόμενο ψήφισμα είναι ένα από αυτά που τάσσονται κατά της αυξανόμενης βίας και της ε, αδικίας. Εγώ αρχικά ε, καλωσόρισα την ε, έρευνα από πλευρά του Διεθνού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα που έλαβαν χώρα κατά τον πόλεμο τη Ανεξαρτησία. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι ο στόχο μα πρέπει να είναι μόνο να τιμωρηθούν οι υπέτη. Η ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει ένα συμφίλιο πόλεμο όπου μόνο ένα μέρο, μόνο μία πλευρά μπορεί να είναι υπεύθυνη για τα εγκλήματα είναι κάτι το πρωτοφανέ στην ιστορία. Θα πρέπει να βρούμε την πραγματική ιστορία, την πραγματική εικόνα. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμού, αλλά η θανατική ποινή είναι κάτι το παράδεκτο. Θα πρέπει να βρούμε την αλήθεια για το τι συνέβη τότε και να δώσουμε ικανοποίηση στα θύματα. Ανταυτού όμως βλέπουμε να αυξάνεται η βία και στην τσεχική δημοκρατία προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για το πώς θα πρέπει να αντιπιστούν οι τιμένοι. Αλλά οι εμπειρίες ε, καταδεικνύουν ότι η καλύτερη λύση ήταν στην Νότια Αφρική γιατί ε, μετά την λήξη των εχθροπραξιών ε, δόθηκε ένα τέλος. Ευχαριστώ. Ε, Τώρα η συνάδελφο Μπασέσκου, αφού ολοκληρώθηκε ο γύρο των από τι ομάδε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια το Μπαγκλαντές ε, έχει μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη με μεγάλες εισαγωγές και πολλέ αλλαδαπέ επενδύσει. Βέβαια η εσωτερική κατάσταση είναι δύσκολη γιατί μέχρι στιγμή ε, σχεδόν μισό πληθυσμό διαβεί κάτω από το όριο τη φτώχεια. Η οικονομική άλλωστε ανάπτυξη απειλείται από τις βίε διαδηλώσει που έλαβαν χώρα το τελευταίο καιρό. Οι μπαγκλατεσιανές αρχές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επανάληψη του διαλόγου με την αντιπολίτευση για να εκτονωθεί η κρίση. Επίσης, οι διαδηλώσεις του Εθνικιστικού Κόμματος έχουν ε, Εξήνεται την κατάσταση, κάτι που αποβαίνει τελικά εις βάρος του μπαγκλατεσιανού λαού. Ευχαριστώ. Περνάμε στο Catch the Eye τώρα. Επειδή είναι πολύ πιεσμένο το χρονοδιάγραμμα, για το Catch the Eye προβλέπονται μόνο δύο ομιλητέ. Ε, θα επιτρέψω να πάρουν το λόγο τρει ομιλητέ και μετά, όσο δεν πήραν το λόγο σε αυτή τη φάση, θα πάρουν το λόγο στι επόμενε συζητήσει. Η συνάδελφος Χουμπνερ, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όταν μιλούμε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Παγκλατές, θα πρέπει να σκεφτούμε και τα, τη 14χρονη Θιάννα Κάτερα. Ε, έχουμε τις α, ε, τραγικές περιστάσεις α, ε, του θανάτου μετά από αποτρόπες α, συνθήκες. Δεν έχουν τέτοια επεισόδια θέση σε ένα πολιτισμένο κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε γιατί συνέβησαν όλα αυτά σε μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι ε, δημοκρατική και αρκετά μετριοπαθής. Τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά δείχνουν ότι στην επαρχία του Μπαγκλαντές και στις μικρές πόλεις και κομοπόλεις όπου δεν λειτουργούν τα δικαστήρια και ουσιαστικά είναι απρόσιτη η παιδεία, αυτό που επικρατεί και πριτανεύει είναι το στιγνό δίκαιο της Σαρία. Ε, έχει τεράστια προβλήματα με την τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η περίπτωση της Χένε Κάτερ δεν είναι δυστυχώς ε, απομονωμένη. Θα ήθελα να απευθύνουμε έκκληση προς την κυβέρνηση για σωστή δράση, για τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την επαναφορά στο κράτος δικαίου, γιατί ήταν κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων της Χένα Κάτερ, αυτής της 14χρονης κοπέλας του Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε στην Χούπνερ και τώρα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πολύ σύντομα με αυτή την ευκαιρία να θυμίσω μία από τις μεγάλες τραγωδίες της ιστορίας του προηγούμενου ε, αιώνα, δηλαδή τον διαχωρισμό ανάμεσα στο Ανατολικό και το Δυτικό Πακιστάν και τη δημιουργία του Μπαγκλαντάς και θα ήθελα εδώ στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου να κάνω μια έκκληση στην κοινωνία του Μπαγκλαντές και στο θεσμούς του Μπαγκλαντές μέσω του δικαστηρίου να μπορέσουν να, κάνουν, να συμφιλιώσουν τη χώρα μέσα στην ε, μεγάλη παράδοση του πολιτισμού του Μπεγγάλη, ε, της, ε, όπως της Βεγγάλης μέσα και από το ποίηματα των διαφόρων ποιητών που συμμετείχαν στο πόλεμο του Μπαγκλατές να σεβαστούν και να ζήσουν σύμφωνα με την μνήμη των διάσημων ε, προγόνων τους, ώστε να επικρατήσει ειρήνη στην χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν έτσι η διαδικασία ΚΑΣΔΙΑ και θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Δαμανάκη. Μικρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, καλωσορίζουμε την υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο του ψηφίσματο σε σχέση με την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαγκλαντέ. Το πρόσφατο κύμα βία που ε, άφησε περίπου 100 νεκρού και πολλού περισσότερου τραυματίε ε, μα ανησυχεί. Η Πατή Εκπρόσωπο, Αντιπρόεδρο Άστον, εξέδωσε δήλωση στις 2 Μαρτίου εκφράζοντας ε, την, ε, την ε, λύπη της για την απώλεια ζώων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Μπαγκλαντές Πρόκειται για μια χώρα με υπερπληθυσμό, με κρέα φτώχεια, ε, περιορισμένους φυσικούς πόρους, ε, προβλήματα στην ασφάλεια τροφίμων, το χαρακτήρα όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, αλλά και θέματα ε, μειονοτήτων. Σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού εξακολουθεί να ζει κάτω από την... το όριο της φτώχεια. Η ανισότητα παραμένει πολύ σημαντικό πρόβλημα, καθώ και η αγραμματοσύνη και η κακή διατροφή. Ε, αυτή η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί στο μέλλον λόγω των κλιματικών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μακρά παράδοση συνεργασίας με τον Μπαγκλαντές για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων εν ώψη των ε, μακρών ε, αντιπαραθέσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις μετά από τις δίκες για τα εγκλήματα πολέμου υπάρχει κίνδυνος να εντατικοποιηθεί η βία, να ενταθεί η βία. Καθώς επιπλέον πλησιάζουν οι κοινοβουλευτικές εκλογές προβλέπονται για το Δεκέμβριο 2013 είτε στις αρχές του Ιανουαρίου του 2014. Ειρηνικέ και καθολικές κοινοβουλευτικές εκλογές θα είναι κλειδί για την ε, δρέωση της δημοκρατίας στον Μπαγκλαντές. Είναι πολύ βασικό οι πολιτικές δυνάμεις να βρουν συνένεση για τον τρόπο ε, διεξαγωγής των εκλογών. Δεν είναι θέμα της διεθνούς κοινότητας να αποφασίσει τη διαδικασία των εκλογών. Εμείς μόνο υποστήριξη μπορούμε να προσφέρουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε τις περασμένες γενικές εκλογές και είναι έτοιμη και να το πράξει και τώρα εάν λάβει σχετική πρόσκληση το, η, ολοκλήρωση των ε, δικών περί εγκλημάτων πολέμου θα επηρεάσουν ε, την κατάσταση. Το γεγονός ότι είμαστε αντίθετοι στη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση και ακόμα και στις περιπτώσεις των χειρότερων εγκλημάτων δεν σημαίνει πως ε, είμαστε υπερασπιστές της ατιμορρησίας. Γνωρίζουμε τα φρικτά γεγονότα που έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1971, τις ε, πολλές ζωές που χάθηκαν και αναγνωρίζουμε τη σημασία της απόδοσης δικαιοσύνης για το λαό του Μπαγκλατές. Έχουμε καλέσει τους ε, εμπλεκόμενους φορείς να δείξουν εγκράτεια και είναι σημαντικό οι μειονότητε να έχουν ειδική προστασία. Χρειάζονται προσπάθειες για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Επιτροπέ ε, Δαμανάκη. Και στο τέλος ε, μας κρατέθηκαν έξι ψηφίσματα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και αργότερα θα λάβουν χώρα οι ψηφοφορίε. Επόμενο θέμα είναι η δραματική κατάσταση των μηνωτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων στο Ιράκ. Καταρχά το λόγο έχουν οι εισηγητές. Ο κύριος ε, Λίζετ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η κατάσταση στο Ιράκ ε, τα τελευταία δεκαετία είναι πολύ περίπλοκη Είχαμε συγκρούσεις και εσωτερικές και εξωτερικές